Per Σας παρακαλώ συνάδελφοι αν θέλετε να καθίσετε. Αρχίζουμε τώρα ε, τη δημόσια συνεδρίαση. Σα Σας παρακαλώ να καθίσετε και να φύγετε από την αίθουσα εάν θέλετε να συνεχίσετε τις κατηδίαν συνομιλίες σας. Συμφωνήσαμε συνάδελφο Λοκ Μπίλερ, που θα προοδρεύσει τις δημόσιες συνεδρίες με τους εμπειρογνώμονες για το θέμα στο Ιράν. Έχουμε την έκθεση πρωτοβουλίας του συναδέλφου Μπέλντερ ε, και ε, να δώσω το λόγο στη συνάδελφο για να προεδρεύσει τη συνεδρία τη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και σας και τους συναδέλφους και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες εδώ πέρα στην ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το Ιράν από μετά τις εκλογές ε, πέρσι τον Ιούνιο ασχολούμαστε πολύ έντονα με την κατάσταση εντός του Ιράν, με την ε, καταπίεση δι... ειρηνικών διαδηλώσεων, ε, με τις συνεχόμενους περιορισμούς οποιασδήποτε κριτικής και είχαμε βεβαίω και το σχετικό ψήφισμα το ΔΕ ε, τον Οκτώβριο ε, φάνηκε σύμφωνα και με την ε, Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας πως υπάρχει κάποια πρόοδος. Οπότε δυστυχώς όμως βλέπουμε πως δεν έχουν υπάρξει επιτυχίες μέσω της διαπραγματευτικής οδού για κάποια αλλαγή. Αντιθέτως διαπιστώνουμε πως ε, υπάρχει μυστική ε, ανάπτυξη καθώς προέκυψε ε, πως γίνεται μυστικός εμπλουτισμός του ουρανίου στο εσωτερικό της χώρας και πρέπει να δούμε το εάν θα οδηγηθούμε σε περαιτέρω κυρίως ακριβώς επειδή δεν υπάρχει καμία πρόοδος όσον αφορά τα πυρηνικά. Τον 2 Φεβρουάριο είχαμε και ένα δεύτερο ψήφισμα που εγκρίναμε για το Ιράν που αφορά και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και τις αποτυχημένες λίγο πολύ προσπάθειες εξέβρεσης πολιτικής λύσης στο ζήτημα το πυρηνικό, οπότε είναι πάρα πολύ θετικό το να κάνουμε αυτή την ακρόαση εδώ πέρα, γιατί όπως είπε ο πρόεδρος ε, πρέπει να προετοιμάσουμε αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας για το Ιράν, αλλά οπωσδήποτε υπάρχει και αυτή η διεθνής συζήτηση περί ε, κυρώσεων σε διεθνές επίπεδο, την οποία πρέπει να κάνουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καλώς ορίζω λοιπόν τους εμπειρογνώμονές μας εδώ πέρα. Θα σας τους παρουσιάσω και σας παρακαλέσω να κάνετε τις δηλώσεις σας. Πρώτα απ' όλα καλωσορίζω τον δόκτορα Πόσο, ο οποίος είναι ερευνητικό συνεργάτης του Ινστιτούτου Επιστήμης και Πολιτικής στο Βερολίνο για τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Ο τομέας ειδικότητας του είναι η εσωτερική και εξωτερική πολιτική της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, η πολιτική άμυνας και ασφάλειας, το πολιτικό σύστημα και οι ε, ευρωιρανικές σχέσεις. Αυτή τη στιγμή δίνει βάρος στην ανάλυση της διαδικασίας μετασχηματισμού των νεοφονταμενταλιστών. Καλώς ήρθατε λοιπόν Καλωσορίζω την καθηγήτρια επίσης Φίρουζε Ναχαβάντη που διδάσκει εδώ πέρα στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών ειδική για την ε, κοινωνικοπολιτική κατάσταση μουσουλμανικών αλλά μη αραβικών ε, χωρών. Έχει πάρα πολλές σχετικές δημοσιεύσεις. Χαίρομαι που σας καλωσορίζω κυρία Ναχαβάντι ακόμη μια φορά ήσασταν και εμπειρογνώμονα στην αντιπροσωπεία του Ιράν. Το ίδιο ισχύει και για τον επόμενο εμπειρογνώμονα, τον κύριο Ρούσμπε, τον δόκτορα Ρούσμπε Πάρση, ο οποίος ε, είναι ερευνητής στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο μελετών ασφαλείας στο Παρίσι και διδάσκει στην Ευρώπη και στη ΣΥΠΑ και έχει πολλές δημοσιεύσεις. Σας καλωσορίζω και θα ήθελα τον να δώσω λόγο στον κύριο Πώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, προσπάθησα να κάνω μία σύντομη επισκόπηση της ιστορικής κατάστασης στο Ιράν και να σας πω, όσον αφορά το, κίνημα αυτό, ε, τα βασικά του στοιχεία ε, είναι ε, ότι είναι η βασική δύναμη αντιπολίτευσης στα πλαίσια του Ισλαμικού καθεστώτος Πρόκειται ε, για διάφορα ε, μικρότερα κόμματα, του οπαδού των κομμάτων αυτών. Πέραν τούτου όμω έχουν έρθει ε, και ομάδε τη κοινωνία των πολιτών όπω το γυναικείο κίνημα και το κίνημα για την ελευθερία. Όμω, αυτά τα κόμματα που εκπροσωπούν ο Μουσαβίο Καρομπή και οι άλλοι κατά κάποιο τρόπο ε, έχουν συμμετάσχει στην ε, δομή της εξουσίας ε, στο σημερινό καθεστώς. Όμως, να σας πω το εξής. Έχουμε τον, το... τον παλιό συνασπισμό ε... Ε... μεταρρύθμισης που περιλαμβάνει και κοσμικούς, μη θρησκευτικούς, δηλαδή, δημοκράτες, ε... μειονότητες κτλ. Όλοι αυτοί δεν δημιουργούν μεγάλες ανησυχίες ε, ε, και δεν αποτελούν απειλή ε, για το καθεστώς. Αλλά το θέμα είναι ότι τώρα υπάρχει κοινωνική αναταραχή και οδήγησαν σε, στην έκρηξη που όλοι είδαμε τον Ιούνιο του 2009. Τώρα, το modus operandi. Μέχρι στιγμής αυθόρμητες μαζικές διαμαρτυρίες, δηλώσεις των λεγόμενων ηγετών του πράσινου κινήματος όπως ο Χαρουμπή και ο Μουσαβή ε, που δίνουν πλατιές και κατευθυντήριε γραμμές, αλλά, αλλά υπάρχει και μεγάλος βαθμός φαντασίας και πρωτοβουλίας ε, ε, που αναπτύσσουν οι νέοι. Υπάρχει ένα ε, είδος ε, ε, ιδεολογικού προβλήματος. Δηλαδή, για να αποφύγουν την, την άμεση αντιπαράθεση με το καθεστώς, οι οπαδοί και, το, και οι βασικοί προτεργάτες του πράσινου κινήματος ακολουθούν ακολουθούν τα αχνάρια της Ισλαμικής Επανάστασης του 79 για να μην θεωρηθούν ως αντικαταστατικοί κτλ. Πέραν όμως αυτού το βασικό είναι η βαθιά απογοήτευση. Και μέχρι, μέχρι στιγμής ε, υπήρχε μια χαλαρή σύνδεση ε, στο κίνημα αυτό των πρασίνων. Ε, όσον αφορά το κίνημα ε, των, ε, των γυναικών, εδώ υπάρχει μια σύνδεση, αλλά δεν έχουν μεγάλη σχέση με τους αντιπολιτευόμενους εκτός της χώρας η επιτυχία του, του κινήματος κρίνεται ανάλογα με ε, τις επιθυμίες του καθεστώτος. Γιατί τι ήθελε το καθεστώς εδώ και χρόνια. Ήθελε να εκδιώξει τις ε, δυνάμεις αυτές μεταρρύθμισης παρόλο που ήταν πιστές στο καθεστώς. Ο Αχμεντίνετζαν ε, ήταν ε, ιδιαίτερα σαφής ε, στην τελευταία του ομιλία και είπε ότι οποιαδήποτε διαδικασία μεταρρύθμισης ε, απαιτεί θυσίες και επίσης ήταν ε, όταν, ε, για, το, γιατί μιλάει όταν χρησιμοποιεί για μεταρρύθμιση, δηλαδή η Ισλαμική ουτοπία, που σημαίνει ότι πρέπει να αφήσει πίσω το καθεστώ τις δημοκρατικές οδούς, ε, τις δημοκρατικές δομές και να προχωρήσει προς κάτι ιδιαίτερα πολιταρχικό και ουτοπικό και αυτό δημιουργεί ιδιαίτερο φόβο. Και όλα αυτά για τη διάδοση του ε, λόγου του Θεού. Αυτή, αυτό το όραμα, αυτή η άποψη του Προέδρου είναι κάτι το οποίο βρισκόταν σε, ε, στη θέση της μειοψηφία τα τελευταία 30 χρόνια και τώρα αρχίζει να αποκτά, ε, να, να παίρνει την κυρίαρχη μορφή έκφραση του καθεστώτος. Όμως, επειδή είχαμε αυτή την, αραχή, την αναταραχή στους δρόμους, δεν μπορούσε, ε, ακόμα και αν προσπαθούσε το καθεστώς, δεν μπορούσε ε, να ε, κρατήσει για πολύ. Και μάλιστα αναγκάστηκε το καθεστώς να ακολουθήσει μια πιο συμφιλωτική γλώσσα. Και αυτό που προσπαθούν τώρα είναι να κερδίσουν αυτά τα στοιχεία των, των μεταρρυθμιστικών δυνάμεων, να τους πάρουν το μέρος τους και να απομονώσουν αυτές όλες τις διαφωνούσες ομάδες μέσα στο κίνημα των Πρασίνων. Για παράδειγμα, ε, υπήρξε μια πολύ σοβαρή απόπειρα να φύγει η λέξη δημοκρατία από οποιαδήποτε δημόσια συζήτηση στο Ιράν. Και τελικά όμως αναγκάστηκαν να αναφερθούν στο Ιράν ως δημοκρατικό κράτος και δύο φορές μάλιστα χρησιμοποίησε ε, ο ηγέτης τους. Αυτό σε μια δημόσια ομιλία. Κοιτάξτε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δέχεται ε, τις θέσεις του, του, του κινήματος αυτού, αλλά αυτή ε, η αρχική ιδέα του καθεστώτος να γίνει ένα απόλυτα απολυταρχικό καθεστώς και ουτοπικό απέτυχε, διότι έχουμε τώρα το κίνημα αυτό ε, το οποίο πέτυχε σε όλα τα επίπεδα θα έλεγα. Το ερώτημα όμως είναι το κατά πόσο μπορεί, είναι βιώσιμο αυτό το κίνημα. Από τον Ιούνιο 2009 και εξή το καθεστώς ε, με ιδιαίτερη επιθετικό τρόπο ε, προχώρησε σε διώξεις των μελών αυτών των πολιτικών ομάδων και των οργανώσεων που ήταν νόμιμες όμως. Που μάλιστα θα έλεγα ότι είναι Ισλαμιστικές οργανώσεις όπως το κόμμα των Μητοχετήν της Ισλαμικής Επανάστασης και το μέτωπο συμμετοχής. Τα στελέχη τους αντιμετώπισαν ε, σκληρές διώξεις με στόχο να παρεμποδιστεί οποιαδήποτε ε, εξάπλωση των οργανώσεων αυτών σε ολόκληρη τη χώρα. Κάτι άλλο τώρα. με εξαίρεση περιστασιακών δηλώσεων των λεγόμενων ηγετών που εκπροσωπούν όμως τα, τα δικά τους κόμματα, δεν υπάρχει σαφής, σαφές συνεκτικό πολιτικό πλαίσιο δράσης. Το καθεστώς δηλαδή μέχρι στιγμής κατάφερε να ε, σταματήσει την έκρηξη ε, αυτή ε, της αναταραχής και, και, την, ε, και να παρεμποδίσει την έκφραση σαφών πολιτικών μηνυμάτων. Άρα, εν συντομία, μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να δούμε μία φάση θριάμβου του καθεστώτος της προσεχής ε, ε, ε, του κινήματος, αλλά αυτή η νίκη θα είναι πύριος νίκη. Γιατί δεν πρόκειται η απογοήτευση να φύγει και σιγά σιγά θα αρχίσει πάλι να, να φουντώνει αυτή η έκρηξη. Ταυτόχρονα η κοινωνική κατάσταση, η κοινωνική αναταραχή ε, και η κατάσταση φτώχειας θα αυξάνονται και θα αυξάνουν και το επίπεδο απογοήτευσης. Άρα λοιπόν μπορούμε να περιμένουμε ε, μια ανασύσταση του κινήματος των πρασίνων και συνέχιση των πολιτικών τους και μέσα στους προσεχείς μήνες. Ο βασικός στόχος του καθεστώτος είναι σαφώς να κερδίσει τους ηγέτες των ε, νόμιμων ακόμα κομμάτων ε, προς το δικό του στρατόπεδο. Όμως θα συνεχιστεί το αδιέξοδο. Δεν πρόκειται να συμβεί αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο και σε επίπεδο αντιπολίτευση αλλά και μέσα στο ίδιο το καθεστώ. Γιατί από τη μια έχουμε του μεταρρυθμιστέ και από την άλλη του μη μεταρρυθμιστέ. Και μέσα στο στρατόπεδο αυτών που θα μπορούσαμε να πούμε των νέων φονταμενταλιστών ή των μη μεταρρυθμιστών αυτή η αυτό το διέξοδο ε, θα συνεχίσει για, καιρό, γιατί φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ρήγμα σε οποιοδήποτε μέτωπο. Και ε, νομίζω ότι τα θέματα, όχι μόνο, τα πράγματα όχι μόνο δεν οδηγούν σε συμφιλίωση, αλλά και σε περαιτέρω επιδείνωση. Ε, Ευχαριστώ η καθηγήτρια κυρία Ναχαβάντη. Σας ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Δέκα λεπτά δεν είναι πολύ χρόνο, άρα θα διαρθρώσω την ομιλία μου σε τρία τμήματα και θα προσπαθήσω να τονίσω σε αυτό που μου φαίνεται το ουσιώδες ε, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στο Ιράν. Θα προσπαθήσω λοιπόν να θέσω πρώτα απ' όλα τα γενικά πλαίσια, στη συνέχεια να αναφερθώ σε κάποια σημεία ε, που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τέλος να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ε, ιδιαίτερα εμείς, ε, ε, τι μπορεί να γίνει μάλλον σε επίπεδο Ευρώπης. Πρώτα απ' όλα να τονίσω ορισμένα στοιχεία τα οποία κατά την άποψή μου είναι σημαντικά για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε ακριβώς πιστεύω ότι πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία στο Ιράν, όπως άλλωστε και η Κίνα, κατά κάποιο τρόπο και σε κάποιο βαθμό, ε, αποτελούν μέρος των δύο, είναι από τις δύο χώρες που έχουν τη χειρότερη βαθμολογία θα έλεγα όσον αφορά ε, τις, ε, ε, ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχουν λοιπόν ένα κοινό στοιχείο και ένα σημείο προσέγγιση οι δύο χώρες αυτές. Δεύτερον, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Κάτι άλλο το οποίο είναι σημαντικό. Ίσως πιστεύω ότι σήμερα έχουμε την τάση να ξεχνάμε ότι όταν μιλάμε με το Ιράν βρισκόμαστε σε μια Ισλαμική δημοκρατία. Η Ισλαμική δημοκρατία τι σημαίνει. Σημαίνει κατά κάποιο τρόπο ότι και, με, και σαφώς θεοκρατικό καθεστώς. Και αυτό αποτελεί ε, τον ακρογόνιο λίθο αυτής της χώρας και το Σύνταγμα από το 79. Όταν μιλάμε για θεοκρατικό καθεστώς, μιλάμε για ένα καθεστώς το, στο οποίο ε, κυρίαρχος είναι ο Θεός και όχι ο λαός. Παρόλο που υπάρχουν μία σειρά από στοιχεία μέσα στο Σύνταγμα τα οποία μιλούν για ε, το λαό. Όταν λοιπόν συζητάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αυτό το στοιχείο της ε, κυριαρχίας του Θεού ε, ε, δεν θα πρέπει να το λησμονάμε ποτέ, γιατί μερικέ φορές έχουμε την τάση να το πράττουμε. Πρόκειται λοιπόν για ένα σύνταγμα το οποίο δημιουργήθηκε μετά από δημοψήφισμα το οποίο οργανώθηκε και αυτό το θεοκρατικό καθεστώς καθιστά κάθε Ιρανό ε, ανήλικο αν θέλετε ενώπιον της εξουσίας. Ο ανώτατος άρχον έχει την, ε, την, την, ε, είναι ο μόνος που έχει δυνατότητα λήψη αποφάσεων. Και μην το ξεχνάμε. Όταν λοιπόν εξετάζουμε το Σύνταγμα, τα διάφορα τμήματα του Συντάγματος, θα δούμε ότι υπάρχουν όλες οι μορφές αντίφασης. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται στο Ιράν. Γιατί? έχουμε και το α και το αντιθετό. από τη μια αναφέρεται η ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα και από την άλλη ε, αναφέρεται ότι οι γυναίκες είναι κατώτερες των ανδρών. Όλα αυτά δεν είναι επινοήματα, ε, δεν είναι υποθέσεις, είναι αντικειμενική πραγματικότητα και μπορούν να επαληθευτούν. Τώρα, το τούλεξέτος, νομίζω ότι όσον αφορά το Ιράν, ε, ίσως γίνονται πολλές εικασίες που δεν είναι βάσιμες. Επανέρχομαι στο θεοκρατικό καθεστώς και στην κατάσταση στο Ιράν σήμερα. Αυτό το καθεστώς και ήδη νομίζω ότι εν μέρη αναφέρθηκε δεν, ε, ε, δεν μπορεί ε, ε, δεν έχει κανένα πρόβλημα όσον αφορά το να υπερασπίσει το καθεστώ αυτό. Θεωρεί ότι έχει δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό το καθεστώ και κάθε δικαίωμα. Κάτι άλλο που είναι χαρακτηριστικό. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ε, επιστροφής των λόγων του 79. Ε, επαναστατικός λόγος, λόγος ε, ε, ε, που αναφέρεται στον τρίτο κόσμο και εδώ είναι ενδιαφέρον να δούμε τη σχέση που έχει σήμερα το Ιράν με άλλες χώρες, ιδιαίτερα του τρίτου κόσμου και να δούμε ποια είναι η επιτυχία της χώρας αυτής. Γιατί και αυτό θα πρέπει να μην το ξεχνάμε και να το τονίζουμε. Αυτά είναι τα πλαίσια μέσα στα οποία θα πρέπει να προχωρήσουμε τον προβληματισμό μας. Τώρα δεν θέλω να επαναλάβω όλα αυτά τα οποία ήδη ελέγχθησαν σε θέματα ε, παραβίασης κάθε είδους κατάφορη παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και μια αρνητική εξέλιξη προς την κατεύθυνση αυτή όπου αυξάνεται ε, με γεωμετρική πρόοδο η βία. Και η καταστολή βεβαίως δεν είναι κάτι το καινούργιο στο Ιράν. Όσον αφορά λοιπόν ε, παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαχωρισμού στα πανεπιστήμια, στην ένταξη στην εργασία, διαχωρισμού ε, ανάμεσα ε, στα δύο φύλλα, διαχωρισμού των ανδρών από τις γυναίκες, ε, το γεγονός ότι, ο, ότι όλες οι μειονότητες αποτελούν αντικείμενο ελέγχου, διωγμού, κακομεταχείρισης, είτε πρόκειται για τις γυναίκες, για τους ομοφιλόφιλους, για τους ανήλικους, ο αριθμός των εκτελέσεων των ετησίων εκτελέσεων στο Ιράν και ιδιαίτερα εκτελέσεων ανηλίκων, πραγματικά όλα αυτά είναι στοιχεία που Όλοι μας τα γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν, σε αυτό το καθεστώς υπάρχει μια ολόκληρη σειρά από αντιπολιτευτικές κινήσεις και εντάσεων που στα πλαίσια αυτά δεν μπορούν να εκφραστούν. Δηλαδή έχουμε μια αντίφαση. Από τη μια έχουμε ένα καθεστώς το οποίο ε, δεν μπορεί να ξεπεράσει τις ε, ε, παροχημένες ιδέες του και μην ξεχνάμε ότι ε, η πλειονότητα του πληθυσμού είναι νέοι. Οι νέοι που κατεβαίνουν σήμερα στους δρόμους δεν έχουν γνωρίσει τίποτα άλλο παρά μόνο την Ισλαμική Δημοκρατία. Και όλα αυτά είναι ενδιαφέροντα στοιχεία και θα πρέπει να το προσέξουμε. Υπάρχει δηλαδή ε, μια, από τη μια έχουμε την ιδεολογία ε, ε, του ότι, ε, ε, την, της ένταξης στην κοινότητα και της ατομικής ιδεολογίας, ιδεολογία ανάμεσα στις πόλεις και στην Ήπεθρο, η νεολαία που ζητά ελευθερία, το θέμα είναι τι είδους ελευθερία ζητά. Ελευθερία για κατανάλωση ή πολιτική κατανάλωση, ή για πολιτική ελευθερία μιλάμε. Εδώ είναι το ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Άρα λοιπόν, στα πλαίσια αυτά, τα οποία σας περιέγραψα, εν συντομία, τι μπορούμε να κάνουμε, ε, νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε από τη μεριά της Ευρώπης, που θα πρέπει να, να ρυθμιστεί απόλυτα, έτσι ώστε να είναι αξιόπιστος ο λόγος της Ευρώπης, είναι να αποφύγουμε τη διπλή γλώσσα. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από αυτό και δεν υπάρχει τίποτα ε, χειρότερο από τη διπλή γλώσσα ε, που να βλάπτει την εικόνα της Ευρώπης έναντι του Ιράν. Δηλαδή από τη μια η Ευρώπη να μιλά για ανθρώπινα δικαιώματα, να μιλά για κυρώσεις, να μιλά ε, για όλα αυτά που γίνονται στο Ιράν και ταυτόχρονα να υπάρχουν ιδιαίτερα επικερδείς συνάψεις, συμβάσεις με το Ιράν. Κοιτάξτε, ε, δεν έχω κανένα πρόβλημα να τα αναφέρω όλα αυτά, διότι ο, ε, ο τύπος ε, έχει αναφέρει κατά κόρον τις συμβάσεις αυτές. Και μιλώ για ευρωπαϊκές χώρες, να μην σας πω τι έχει γραφτεί για τους Αμερικανούς που και αυτοί έχουν επενδύσει ιδιαίτερα στη χώρα αυτή. Σήμερα, αυτή την εβδομάδα ε, αναφέρθηκε πάνω από δις ε, ε, δολάρια είναι οι επενδύσει των Αμερικανών στο Ιράν. Άρα λοιπόν αυτό ε, αμαυρώνει ιδιαίτερα την αξιοπιστία. Πώς θέλετε να περάσετε ένα αξιόπιστο μήνυμα εφόσον οι πολιτικοί στην Ευρώπη δεν μπορούν να ελέγξουν, να ελέγξουν το οικονομικό σκέλος. Πώς θέλουν λοιπόν να ελέγξουν τον κόσμο. Καταλαβαίνετε αυτό είναι το ερώτημα. Και αυτό είναι πραγματικά το στοιχείο που κατά την άποψή μου είναι κεντρική σημασία. Δηλαδή, ποιε είναι οι προτεραιότητε τη Ευρώπη. Το να μιλάμε για αξίε ε, και για προάσπιση οικονομία. Μερικέ φορέ αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Δεύτερο στοιχείο, ε, νομίζω ότι έχω ξεμπίσει το χρόνο μου και θα είμαι πολύ γρήγορη. Πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι ε, αναφέρουν οι Ιρανοί. Γιατί πιστεύω ότι εδώ δεν έχει γίνει κατανοητό στην Ευρώπη το τι θέλουν να πούν οι Ιρανοί. Δεν μιλώ να ε, τους δικαιολογήσουμε, αλλά τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να τους καταλάβουμε. Όσον αφορά τώρα τις κυρώσεις, ε, δεν έχω το χρόνο λοιπόν να αναφερθώ στο ζήτημα αυτό, αλλά ο τρόπος με τον οποίο γίνονται, εδώ ε, είναι διάλογος κουφών. Ε, είναι κουφό το κράτος του Ιράν που δεν, που δεν θέλει να ακούσει αυτά που του λένε οι υπόλοιποι. Όλα όσα που θέλει να αντιλήσει τα διδάγματα. Νομίζω λοιπόν ότι σε σχέση με αυτά τα οποία γίνονται σήμερα στο Ιράν, ε, λαμβάνοντα υπόψη ότι έχουμε ένα κουφό κράτο, με το οποίο ε, όμω συνεργαζόμαστε σε οικονομική βάση, καταλαβαίνετε ότι τουλάχιστον πρέπει να προσπαθήσουμε να υποστηρίξουμε τον πληθυσμό της χώρας και να το καταλάβουμε, τον ακούσουμε. Και τέλος, όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα, πιστεύω ότι ίσως για να καταλάβουμε τι γίνεται, θα έπρεπε να κάνουμε ένα παραλληλισμό με την κρίση των πυράβλων στην Κούβα το 1963. Νομίζω ότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να καταλάβουμε ποιες είναι ενδεχομένως οι προθέσεις. Ίσως μια άλλη ερμηνεία, παρόλο που δεν μπορεί να αρνηθεί ότι οι Ιρανοί κάνουν, αρκετά, κάνουν τεράστια πράγματα προς την κατεύθυνση αυτή. Ίσως λοιπόν πάρα πολλά πράγματα. Ίσως λοιπόν, ε, αν δούμε το θέμα από τη σκοπιά αυτή, θα μπορέσουμε να καταλάβουμε και με διαφορετικό τρόπο τα κίνητρά τους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κυρία Ναχαβάντη. Τώρα θα δώσω τον λόγο στον Δόκτωρα Πάρση, παρακαλώ. Ευχαριστώ, καλημέρα. Μου ζήτησαν να μιλήσω για τις ε, περιφερειακές ε, πτυχές και θα το κάνω αυτό και μετά ως τελευταίο θα εκμεταλλευτώ τη θέση μου για να αναφερθώ στα ζητήματα που αναφέρθηκαν και οι συνάδελφοι όσον αφορά λοιπόν την περιοχή εκεί πέρα. Μία από τις βασικές ελλείψεις που βλέπουμε συνεχώς είναι η έλλειψη ενός κοινού πλαισίου ασφαλείας. Δηλαδή, αν δούμε τη Μέση Ανατολή, ειδικά τον Περσικό κόλπο, βλέπουμε πως οι χώρες εκεί πέρα έχουν θέσεις αμφιταλαβευντευόμενες έναντι του Ιράν. Απ' την άλλη υπάρχει ιστορική αντιπαλότητα και φόβος του μεγαλύτερου γείτονα εκεί πέρα στην περιοχή, ανεξαρτήτως του πυρηνικού ζητήματος, από την άλλη, ως μόνιμοι γείτονες, γνωρίζουν τις επιπτώσεις, τις καταστροφικές, εάν ε, οδηγηθεί η κατάσταση σε ένοπλη σύγκρουση. Οπότε, εάν δούμε την νότια όχθη του Περσικού κόλπου, από τη μία θέλουν το πυρηνικό πρόγραμμα να είναι μόνο πολιτικό και υπό αυστηρές εγγυήσεις, από την άλλη δεν φαίνεται να έχουν όρεξη για ένα συνεχόμενο πόκερ όπου τα στοιχήματα συνεχώς θα ανεβαίνουν και μοιραία θα οδηγηθούμε σε ενόπλη σύγκρουση. Και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε όταν συζητάμε το τι θα είναι γείτονε. Τώρα υπάρχουν πολλές χώρες στην νότια ακτή που έχουν καλές σχέσεις όπως το Κατάρ και εμπορικές και άλλες Μία από τις πιο σημαντικές διεξόδους, π.χ. οικονομικές είναι το Ντουμπάι και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Υπάρχουν κοινέ ε, ανησυχίες και αμοιβαίοι, αν θέλετε, φόβοι και ένας από αυτούς είναι η εθνοτική και θρησκευτική πτυχή. Δηλαδή το Ιράν πάντα φοβάται πως οι άλλοι θα προσπαθήσουν να το διχάσουν σε θρησκευτικές γραμμές, ειδικά στα Ανατολικά, στο Βαλουχιστάν με το Πακιστάν και στις χώρες του Περσικού κόλπου υπάρχει φόβος των σιητικών μειονοτήτων που μπορεί να ενθαρρυνθούν από την κυβέρνηση της Τεχεράνης. Από αυτή την έννοια φαίνεται πως φοβά το Γιάννη στο θεριό και το θεριό το Γιάννη και προσπαθούν όλοι να μην υποκύψουν σε αυτόν τον πειρασμό αλλά οι κατηγορίες εκτοξεύονται κατέρασταν. Και δεν ξέρω αν υπάρχει βάση πίσω από αυτές τις κατηγορίες τώρα για να επανέλθουμε σε αυτή την προσέγγιση του κοινού πλαισίου ασφαλείας. Όλοι το βλέπουν ότι ό,τι κερδίσουν θα χάσει ο άλλος. Έτσι το βλέπουν οι ΙΠΑ, έτσι το βλέπουν στη Μέση Ανατολή. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι ταυτόχρονα ενώ οι γειτονικέ χώρες του Ιράν δεν θα σύγκρουση, φοβούνται μια προσέγγιση Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών που θα τις αφήσει έξω από το παιχνίδι. Οπότε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα λύσης της υπόθεσης αυτής από συμβατική σκοπιά είναι πως δεν μπορούν να φανταστούν μια συνύπαρξη η οποία δεν θα βασίζεται στην αποτροπή. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Τώρα, θα ήθελα να επανέλθω σε κάποια ζητήματα που ανέφεραν και οι συνάδελφοί μου και ειδικά όταν μιλάμε για κυρώσεις. Ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να ρωτηθούμε όταν μιλάμε για περαιτέρω κυρώσεις είναι, κυρώσεις είναι τι θέμα να επιτύχουν οι κυρώσεις στο ΙΕ αφορούν συγκεκριμένα τα πυρηνικά. Οπότε ορισμού είναι στοχευμένες. Γιατί ο στόχος είναι πολύ συγκεκριμένος. Τώρα, κάποιες χώρες, π.χ. είπα, είχαν, έχουν ε, επί 30 χρόνια επιβάλει κυρώσεις στο Ιράν. Εγώ δεν ε, βλέπω τι έχουν επιτύχει. Η δε ιδέα των περαιτέρω κυρώσεων κατά του Ιράν βασίζεται στο ότι υπάρχει κάποιος συγκεκριμένο στόχος που μπορεί να επιτευχθεί εντός του Ιράν που με τη σειρά του θα επηρεάσει το πυρηνικό ζήτημα ή ακόμη παραπέρα το ίδιο το καθεστώς. Τώρα, οι κυρώσεις μοιραία θα επηρεάσουν την κοινωνία. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Το ζήτημα λοιπόν είναι πώς νομίζουμε ότι θα αντιδράσει μετά ο Ιρανικός λαός. Οι ε, που βλάπτουν την οικονομία του Ιράν θα τους βλάψουν όλους. Και είναι ρίσκο να πιστεύουμε ότι μόνο την κυβέρνησή τους θα κατηγορήσουν. Σημαντικό είναι επίσης να δούμε το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί το περνικό ζήτημα δεν συζητιέται εντός του Ιράν. Δεν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις εντός του πολιτικού φάσματος του Ιράν για το πυρηνικό ζήτημα. Οπότε αν έχουμε αντίδραση εντός του Ιράν, τότε περισσότερη αντίδραση θα βρούμε με το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και δικαίως και εξορισμού μετά αυτή η συζήτηση δεν απευθύνεται σε μια συγκεκριμένη παράταξη πολιτική. Και αυτό είναι σημαντικό. Εάν δεν θέμε να μπλεχτούμε στην εσωτερική πολιτική της ίδιας της Τεχεράνης, που δεν θα είναι και πολύ παραγωγικό, νομίζω συμφωνούν όλοι. Υπό αυτή την έννοια θα έλεγα πως το πυρηνικό ζήτημα δεν θα αλλάξει στο προσεχές μέλλον. Εκεί που μπορούν να κινηθούν τα πράγματα είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και εκεί μπορούμε να κερδίσουμε σε αξιοπιστία και εντός και για εμάς που είμαστε εκτός του Ιράν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δόκτωρα Πάρση για τις εκτιμήσεις σας και τις προτάσεις σας. Τώρα μπορούμε να συζητήσουμε μέχρι τις 12 και μισή, μετά πρέπει να γίνει ένα διάλειμμα. Έχω πέντε ομιλητές, έξι. Και εδώ θα κλείσει ο κατάλογος των ομιλητών. Θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα ερώτημα προς εσάς κύριε Είπατε και παρατηρήσαμε όλοι πως η κυβέρνηση έμαθε να το πώς μπορεί να διαταράξει την κινητοποίηση του πράσινου κινήματος και με την σύγχρονη τεχνολογία. Είσαστε λοιπόν υπέρ της βοήθειας ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποκτήσουν αυτές οι ομάδε σύγχρονη τεχνολογία για να ξεπεράσουν αυτά τα εμπόδια. Βέβαια, αυτό σημαίνει πως εδώ πέρα θα παραβιαστούν ε, ορισμένες κυρώσει. Λοιπόν, ο κύριο Μπέλτερ πρώτα απ' όλα στον κατάλογο μου. Κύριε Μπέλτερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να συγχαρώ τους ε, εισηγητές, πολύ ενδιαφέροντες. Σύντομα, αναρωτιέμαι Βλέπουμε στο Ιράν αυτή τη στιγμή μια επαναστατική διάθεση, αλλά ταυτόχρονα ο κλήρος έχει διαφορετικές ε, κατευθύνσεις. Υπάρχουν ε, διάφορες δυνατότητες αφενός και προς μια ήπια αντιμετώπιση και υπάρχει μια αντιπολίτευση του κλήρου που μιλάει και για κάποια πιθανότητα διαλόγου αλλά βεβαίως ε, υπάρχει εδώ πέρα και το ζήτημα της ασυριακής, ε, της αραβικής ε, μειονότητας, των βαλούχων, όλοι αυτοί, όλα αυτά που είναι τροτά σημεία του, του καθεστώτος και βεβαίως ε, υπάρχει και σε έναν... Ε, είναι, το καθεστώς ε, έχει εμπλακεί σε ένα ηλεκτρονικό πόλεμο. Θεωρείτε πως θα πρέπει να, εξασφα... να τονίσουμε πως πέρα από τα πυρηνικά ανισχούμε πάρα πολύ και για τα θεμελιώδη δικαιώματα και για την ελευθερία των πολιτών του Ιράν. να υπάρξει όμως μια κάποια τέτοια στήριξη χωρίς να φανεί ότι εμείς παρεμβαίνουμε από το εξωτερικό στην πολιτική του Ιράν. Ευχαριστώ κύριε Μπέλτερ. Να ε, σας υπενθυμίσω όμως να είστε ως το δυνατόν πιο σύντομοι για να μπορέσουν να απαντήσουν και οι δικοί μας. Κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ για μια, εξαιρετική, για μια σειρά από εξαιρετικές παρουσιάσεις. Έχει ενδιαφέρον να δει κανείς ότι αυτό που μας λέτε είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα γιατί αλλιώς δεν θα λυθούν γενικότερα τα προβλήματα με το Ιράν. Μας είχαν προειδοποιήσει ότι δεν μπορούμε να λύσουμε το θέμα το πυρηνικό εις βάρος του προβλήματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το θέμα δεν είναι να βρούμε μόνο λοιπόν τις ευφυείς κυρώσεις, αλλά τι είδους προληπτικά μέτρα μπορούμε να επιλέξουμε έτσι ώστε να βοηθήσουμε την κατάσταση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε τώρα τα Euronews FRC είναι ένα πρώτο μέτρο. Το θέμα δεν είναι μόνο το Ιράν, βέβαια. Έχουμε τους Μουτζαχιντίν Χάλκ από πίσω. Θα ήθελα να μάθω ποια είναι η αξιοπιστία τους και το βάρος τους στο Ιράν. Έχει σημασία για τα μέλη του Κοινοβουλίου να γνωρίζουν ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Ευχαριστώ Γκάλερ. Ναι, δύο σύντομες ερωτήσεις. Η μία φορά τις μειονότητες. Κατά πόσο συμμετέχουν σε αυτό το πράσινο κίνημα. Και ίσως είναι σημαντικό να απομακρυνθεί από αυτή την, το συγκεντρωτισμό το Ιράν για να δούμε τι θα γίνει και με τις ε, μειονότητες για το πώς θα μπορέσει να οικονομηθεί μια πλειοψηφία. Τέλος, για τις κυρώσεις μήπως θεωρείτε πως στοχευμένες κυρώσει κατά προσώπων που έχουν αξιώματα στο καθεστώς. Δηλαδή να μπορούν πλέον να ταξιδέψουν, να παγώσουν οι λογαριασμοί τους. Έχει κάποιο αποτέλεσμα. Αυτές οι χιλιάδες ε, που είναι στα θρησκευτικά ιδρύματα, στη δικαιοσύνη, σε διάφορες ε, θέσεις. Το να τους βάλουμε σε κάποιες λίστες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρώσεων και να τις ε, δημοσιεύσουμε, νομίζω έχει κάποιο αποτέλεσμα. Δηλαδή διαπιστώνεται ότι είναι και συνδεδεμένοι και με το καθεστώς και δεν θα μπορούν να, να αρνηθούν κάτι τέτοιο. Θεωρείτε πως κάτι τέτοιο μπορεί να ασκήσει πίεση στο εσωτερικό. Ευχαριστώ κύριο Σαλάτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μια αρχική σκέψη. Στα πλαίσια της πολιτικής μου εμπειρίας έχω συνηθίσει να χρησιμοποιώ κάποια περίπλοκη γλώσσα, αν θέλετε, βυζαντινού τύπου γλώσσα αλλά πραγματικά οι τρεις ομιλητές σήμερα ξεπέρασαν κάθε δυνατότητα που υπάρχει κανείς σε έμεσο τρόπο έκφρασης. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να μιλήσουμε πιο απλά. Πιστεύετε ότι αυτή η θεοκρατία είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να ισχύσει για τη χώρα αυτή είναι πραγματικά ο τρόπος σκέψης τους αυτός, ενώ ξέρουμε ότι για μας κάτι τέτοιο δεν μπορούμε να το συμμεριστούμε. Αυτοί όμως πραγματικά ένα τέτοιο νόμο, ένα τέτοιο καθεστώς θα το δεχτούν. Μια δεύτερη ερώτηση. Υπάρχει μια υπόθεση η οποία τίθεται για τη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αντιπολίτευση την Ιρανική και όχι μόνο με τις κυβερνητικές δυνάμεις. Τρίτη ερώτηση. Θα συμφωνήσουν οι τρεις εμπειρογνώμονες να ζητήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα πάγωμα των εκτελέσεων τουλάχιστον ώσπου να οργανωθεί ένα ταξίδι δικό μας στη χώρα αυτή. Σας παρακαλώ να είστε πραγματικά σύντομος. Uh, ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους ομιλητές να αναφερθώ και εγώ στις κυρώσεις γιατί φαίνεται πως είναι πολύπλευρες και πολύπλοκες. Δεν έχουμε προσδοκίες για άμεση δράση και αλλαγή στο πυρηνικό πρόγραμμα. Θέλουμε να βελτιώσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και φαίνεται πως η κυρώση είναι η τελευταία λύση για να διασώσουμε και τη δική μας αξιοπρέπεια μετά τις ε, προσβολές ε, που υποστήκαμε με την παραβίαση προθεσμιών κτλ. Αλλά φαίνεται πως ε, είπα... Σταμάτησαν κάποιες κυρώσεις, ειδικά όσον αφορά το λογισμικό για να βελτιωθούν οι επικοινωνίες από τα κάτω προς τα πάνω, παρά το ότι υπήρχαν κάποιες ε, κυρώσει έναντι ατόμων που ήταν κατηγορούμενα για εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητα. Θεωρείτε λοιπόν ότι ίσως και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει κάποια ανάλογα βήματα. Και ο κύριο Λέχνερ, ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομο Η κυρία Ναχαβάντη αναφέρθηκε στι οικονομικές σχέσεις ε, και τι επιχειρήσεις ε, που συναλλάσσονται με το Ιράν και μίλησε για διπλή ηθική. Εντάξει, το αντιλαμβάνομαι. Τώρα, μιλάμε πράγματι και για κυρώσεις. Αυτό είναι η κατάληξη της ε, λογικής μας. Μιλάμε για πλήρη διακοπή των εμπορικών σχέσεων και επανερχόμαστε εδώ πέρα. Αφορά αυτό πλήττει τον πληθυσμό, έχει κανένα θετικό αποτέλεσμα. Θέλω να δω πώς το, πώς το βλέπετε και πώς σχετίζονται αυτά τα δύο μεταξύ τους. Σας ευχαριστώ και τώρα έχετε την, ε, το αδύνατο έργο βέβαια να απαντήσετε σε όλα αυτά. Σας ξεκινήσουμε σας κύριε Ναι. Όσον αφορά... Σχετικά με το διαδίκτυο, οι Ιρανοί έδειξαν πάρα πολύ φαντασία και χρησιμοποίησαν όλα τα σύγχρονα μέσα τα οποία έχουν στη διάθεσή τους, είτε νόμιμα είτε όχι ακριβώς νόμιμα. αν θέλει κανείς να αγοράσει κάποιο λογισμικό ή κάποιο μηχάνημα θα τα βρει εύκολα στην Τεχεράνη. Το καθεστώς έχει βοηθήσει στο να εισαχθεί, εισαχθεί η νέα τεχνολογία στο Ιράν. Τη χρησιμοποιούν εξ αρχής ε, οι αρχές, τη χρησιμοποιούν έξυπνα, παίζουν τον δικό τους κυβερνοπόλεμο, έχουν διάφορες διαδικασίες ελέγχου και μελετούν τις επιπτώσεις του ίντερνετ στην κοινωνία. Υπάρχει λοιπόν μια συζήτηση ενδιαφέρουσα όχι μόνο στο εσωτερικό του κινήματος αλλά και πέραν και δεν φοβούνται να χρησιμοποιούν το ίντερνετ, ε, τη χρήση του ίντερνετ από τον Ιρανικό πληθυσμό ή του καθεστώτος. Παρακολουθούν, ελέγχουν το φάσμα των συχνοτήτων και αυτό είναι απαράδεκτο. Ελέγχουν έτσι και αλλιώς και τις τηλεπικοινωνίες γενικότερα και ε, το διαδίκτυο ελέγχεται επίσης από το καθεστώς. Αυτό το οποίο τους ενδιαφέρει είναι να μην χρησιμοποιηθεί το διαδίκτυο για να οργανωθούν μεγάλες διαδηλώσεις και αυτό επίσης καταφέρνει και το ελέγχει η κυβέρνηση. Ανησυχούν λοιπόν για το δίκτυο αλλά έχουν αναπτύξει παράλληλα και ένα σύνολο μέτρων για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του. Από πλευράς του πληθυσμού υπάρχει το θέμα της πειρατείας στο διαδίκτυο, το οποίο είναι αρκετά διαδεδομένο. Για τις εθνοτικές μειονότητες υπάρχει ιδεολογική θα έλεγα αποστροφή προς την κυβέρνηση και το Ιράν γενικότερα στην περιοχή του Βαλοχιστάν. Τον Οκτώβριο η κυβέρνηση υπέστη εκεί μια πολύ μεγάλη ήττα εκλογική. Πέραν αυτού το καθεστώς του Ιράν είναι ιδιαίτερα ανεκτικό απέναντι στις μειονότητες. Οι μειονότητες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τη γλώσσα τους παρόλα αυτά, αλλά λέει το Σύνταγμα, αλλά δείχνει η πραγματικότητα και βλέπουμε ότι οι Σουνίτες συν κάποιες εθνοτικές μειονότητες, συν κάποια αντιστασιακά κινήματα και οι Κούρδοι πολλές φορές ε, την χάνουν τη φροντίδα σε εισαγωγικά του καθεστώτος. Το Ιρανικό καθεστώς δεν σέβεται λοιπόν μπορούμε να πούμε το Σύνταγμα, όλα τα σημεία του Συντάγματος σχετικά με τις εθνοτικές μειονότητες η επαναστατική φρουρά ενισχύεται, αλλά οι συνάδελφοι ίσως θα αναφερθούν σε αυτό περισσότερο. Όχι, να πω εγώ κάτι γιατί την... Ε, ε, υπάρχουν δύο στοιχεία. Από τη μία, οι ερωμένοι ποτέ δεν ήταν ε, θα έλεγα ενωμένοι πολλές φορές ήταν εναντίον του καθεστώτος και πολλοί θεολόγοι και πολλοί ηγέτες ε, στον τομέα των θεολογικών ήταν εναντίον του καθεστώτος και ε, ασχολούνται με την πολιτική όχι γιατί είναι κληρικοί αλλά γιατί ανήκουν σε συγκεκριμένες πολιτικές παρατάξεις. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα με τους ε, ιερωμένους οι οποίοι έχουν συγκεκριμένες απόψεις και συνδυάζουν την πίστη τους με το πολιτικό Ισλάμ. αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί αγιατολάδες και πάρα πολλοί απλοί κληρικοί στη φυλακή ε, σήμερα. Για διάφορους λόγους ο Σάχης δεν θα τολμούσε ποτέ να το κάνει αυτό. Οι Μπασιτζοί τώρα εκφράζουν ε, τους νέους ιδεολόγους της δεκαετίας του 80 ε, και οι οποίοι τώρα θέλουν και αυτοί το δικό τους κομμάτι από την πίτα. Αυτά για τους Μπασιτζοί. Λυπάμαι, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Κυρία Ναχαβάντη, δεν θα μακρηγορήσω. Να επανέλθω στο θέμα του κλήρου, ότι όχι μόνο ένα μεγάλο τμήμα του κλήρου είναι στη φυλακή αυτή τη στιγμή, διώκονται, είναι κατοίκον περιορισμό, σε κατοίκον περιορισμό, αλλά υπάρχουν ε, συγκεκριμένες κυρώσεις και ειδικά δικαστήρια που αντιμετωπίζουν τα, ε, τα θέματα των κληρικών. Οι κληρικοί λοιπόν υφίστανται την καταστολή με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Και πάντα σχετικά με τον κλήρο υπάρχει μία κάποια ελπίδα θα έλεγα για το αύριο γιατί ένα τμήμα του κλήρου είναι υπέρ του διαχωρισμού της πολιτικής και της θρησκείας. Και αυτό ακριβώς το τμήμα του κλήρου πρέπει να το ενισχύσουμε, να το ακούσουμε και δυστυχώς δεν, κανείς δεν στρέφει ε, ε, τα ότα του προς την κατεύθυνση αυτή. Τώρα για τους Μοτζαϊντίν. Αυτό το οποίο δεν υπάρχει πια σήμερα, τουλάχιστον στο εξωτερικό και ίσως ούτε και στο εσωτερικό, κατά είναι κάποιοι ηγέτες της αντιπολίτευσης. Το είδαμε αυτό στα πλαίσια του πράσινου κινήματος. Δεν νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι εκ των υστέρων διεκδίκησαν την ηγεσία του κινήματος αυτού ήταν πραγματικά σε θέση να το κάνουν ο κύριος Μουσαουή και άλλοι. Και από την άλλη στο εξωτερικό δεν υπάρχει ένας ηγέτης και αυτό είναι η αδυναμία της έκφρασης της Ιρανικής αντιπολίτευσης. Στο Ιράν οι Μουτζαϊντίν δεν αποτελούν μια εναλλακτική λύση. Για πολλούς Ιρανούς είναι χειρότερη από το καθεστώς. Η σύνθεση ιδεών των Μουτζαϊντίν Χάλκ είναι χειρότερη για πολλούς Ιρανούς από ό,τι τα του καθεστώτος. Παρ' όλα αυτά είναι δραστήριοι και επίσης προχωρούν και έχουν παρουσία στην Δύση χωρίς όμως να την χάνουν της ε, στήριξης των Ιρανών για τις μειονότητες. Το θέμα των μειονοτήτων εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει λίγο αποκριβεί θα έλεγα, λόγω του ότι γενικά έχουμε να κάνουμε με Ιρανούς και δεν υπάρχουν εσωτερικές διαφορές ανάμεσα στα διάφορα κόμματα και στους διάφορους πληθυσμούς. Είναι κάτι όμως το οποίο έχει αρχίσει και κλονίζεται υπάρχει μια κάποια αντιπολίτευση, αντίθεση μάλλον, μια κάποια θα έλεγα δυσανεξία ε, κάποιων μειονοτήτων απέναντι στους Πέρσες, στους Ιρανούς, Ιρανούς δηλαδή. Υπάρχει μια δυσθυμία των αραβικών πληθυσμών, των Σουνιτών απέναντι στη σιτική πλειοψηφία, σχετικά με τη θεοκρατία εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει εδώ να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε κάτι περισσότερο. Προσωπικά νομίζω ότι δεν θα πρέπει να αναμειγνύουμε τα πράγματα. Η πολιτική και η θρησκεία δεν κάνουν ζάφτη. Οι Ιρανοί δεν κατάλαβαν πολύ καλά τα πράγματα όταν πήραν μέρος στο δημοψήφισμα για τη θεοκρατία. το να σταματήσουν προσωρινά οι εκτελέσεις, δεν ξέρω γιατί οι Ιρανοί να δεχθούν να σταματήσουν οι εκτελέσεις αυτές προσωρινά, δεν δέχονται καμία συζήτηση γύρω από την ποινή, γιατί δεν θεωρούν ότι οι συνομιλητές τους είναι ιδιαίτερως αξιόπιστοι. Σχετικά με τις κυρώσεις, και θα σταματήσω εδώ, οι κυρώσεις οι οποίες θα θίξουν αυτούς οι οποίοι πραγματικά κατέχουν τον πλούτο στο Ιράν θα ήταν οι πραγματικές θετικές κυρώσεις. Αλλά προς στιγμή αυτό το οποίο βλέπουμε και αυτό που ακούμε από τη Δύση είναι να δημιουργούνται νέοι εχθροί. Να μπλοκάρονται ας πούμε λογαριασμοί Ιρανών στην Ευρώπη. Ε, δεν αποτελούν αυτοί θα έλεγα το καθεστώς προφανώς, ούτε είναι και αυτοί οι οποίοι ασκούν φυσικά την αντιπολίτευση. Ευχαριστώ και τέλος κύριος ο δόκτωρας Πάρση. Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι όσον αφορά το Ιρανικό Σύνταγμα περιέχει ορισμένα σχιζοφρενικά στοιχεία θα έλεγα. Αλλά ακόμα και αυτό, ακόμα και αυτό θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε αν τουλάχιστον ακολουθούσαν το σύνταγμά τους. Υπάρχουν πολλές ελευθερίες στο Ιρανικό Σύνταγμα. Το πρόβλημα είναι όμως ότι ε, το κράτο και η πολιτεία δεν σέβεται το Σύνταγμα. Όσον αφορά τώρα την αντιπολίτευση, εγώ είμαι πιο αισιόδοξο όσον αφορά την ιστορική αντιπολίτευση. Για την εξωτερική θα σα έλεγα ότι οποιοδήποτε αντιπολίτευση βρίσκεται τώρα έξω από τη χώρα έχει αξιοπιστία μόνο εφόσον ευθυγραμμίζεται με την εσωτερική αντιπολίτευση. Ε, οι Μουτζαντινεχάν χάσανε την αξιοπιστία του εδώ και καιρό. Ε, όταν ε, πολέμησαν με το Χουσέιν κατά του Ιράν. Ε, εξεπιστία έχουν μόνο εδώ, για παράδειγμα. Στο, Ιράκ, στο Ιράν δεν έχουν εξεπιστία. Για τις κυρώσεις νομίζω ότι ίσως ε, θα μπορούσε κάποιος ε, να προχωρήσει περαιτέρω και να πούμε ναι, ναι, μπορείτε να να στοχεύσετε συγκεκριμένε ομάδε μέσα στην κυβερνητική δομή όσον αφορά τι κυρώσει. Αλλά ο μακροπρόθεσμο στόχο είναι ε, να, ε, αν θέλετε, να αντιμετωπίσετε τις ριζοσπαστικές ε, άκρες του κράτους και να υπάρξει ένα είδος ομαλοποίησης και εσωτερικό επίπεδο, αλλά και σε σχέση με τους γείτονε, τότε η δέσμευση είναι κάτι το οποίο απαιτείται. Μόνο μία χώρα ξέρουμε στην οποία οι κυρώσεις να άλλαξαν την εσωτερική ε, συμπεριφορά και, και, και κατ' επέκταση και εκτός. Η Νότια Αφρική, αλλά αυτή ήταν η εξαίρεση, όχι ο κανόνας. Άρα το αντεπιχείρημα θα ήταν να δεσμευτεί, ε, να υπάρξει δέσμευση σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα μέτωπα ε, ε, συμμετοχή του Ιράν δηλαδή και όχι να έχουμε την εντύπωση ότι αν το βάλουμε στην άκρη θα είναι πιο συνεργάσιμο γιατί γίνεται αυτή η άκρη ε, δεν είναι στον έλεγχό σας δεν μιλάμε για το 19ο αιώνα όπου το Βρετανικό πολεμικό ναυτικό μπορεί να κάνει αποκλεισμό στη χώρα που δεν της αρέσει γιατί πάντα θα υπάρχει μια Κίνα Ευχαριστώ ναι, Ευχαριστώ και τους τρεις εμπειρογνώμονές μας ε, για τις ε, ενδιαφέρουσες αυτές παρατηρήσεις. Ε, κοιτάω και το ρολόι. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους για την προσοχή σας και εδώ πέρα λύεται η συνεδρίαση.